det och Καλησπέρα σα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Το σημείο 1 στη μέση διάταξη ήταν η συνεδρίαση των συντονιστών. Το αφήνουμε αυτό λοιπόν. Mm. Ε, προχωράμε στην, ε, στο σημείο 2 έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε, οπότε προχωράμε. Ε, είμαστε 10, ε, έχουμε απαρτία. και ναι, αλλιώς δεν θα είχα ξεκινήσει τη συνεδρίαση. θα ξαναμιλήσω σου ναι, ναι, εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Προχωράμε στο σημείο 3. ανακοινώσει του Προέδρου δεν υπάρχουν. Ε, σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει ε, που έλαβαν οι συντονιστέ. Έχετε τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 3 ε, Οκτωβρίου και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε και να αρχιοθετήσουμε τα πρακτικά. Ε, σημείο 5. Just a moment, sorry. Uh, uh, uh, e Έχουμε λοιπόν τον χάρτη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας του φύλου να δώσω το λόγο στην κυρία Κλιβέτη πριν ε, περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ε, απλά θέλω να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα κοινό ψήφισμα για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς όλων των πολιτικών ομάδων. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, ότι πριν ένα χρόνο όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να στηρίξουν το ψήφισμα αυτό που έχω μπροστά μου και το οποίο γνωρίζετε. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε σήμερα λοιπόν αποτελεί συνέχεια της κοινή απόφασης όλων των πολιτικών ομάδων. Κύριε Κλειβέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία και θα μιλήσω αγγλικά. Ξεκινάμε με την τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 11 και 12 είναι όμοιες. Χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην ε, συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29, χωριστή ψηφοφορία σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τέταρτο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, αρχή της ψηφοφορίας. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Okay, we add... And definitely Σαφώς εγκρίνεται. Ε, θα ψηφίσουμε πάντως, θα προσθέσουμε την ε, ψήφο σας. Ε, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Το αποτέλεσμα. 11 ε, στις 12 ψήφους, αλλά έχουμε 12 υπέρ. 12-3. då går vi vidare eh, på dagordningen och... Ωραία, προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Προχωράμε. Παρακαλώ. Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Σούμπερ. Παρακαλώ. Ε, ε, Γεια σας σε όλους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι δεδομένου ότι δεν είχα πολύ χρόνο για να συντάξω την ε, έκθεση μου, έκανα διάφορες επιλογές σε σχέση με την εξέλιξη της ισότητας των δύο φύλων και είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί, αλλά είμαι σίγουρη ότι με την κατάθεση τροπολογιών οι ελλείψεις αυτές θα ξεπεραστούν. Όταν μιλούμε για ισότητα το 2012, χρονιά κατά την οποία είδαμε ότι σε διάφορες χώρες εφαρμόστηκαν μέτρα πολιτικής φύσης ε, εν ώψη της ε, λεγόμενης λιτότητας είδαμε ότι παγιώθηκαν αυτά τα μέτρα και τουλάχιστον σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας οικονομικής κρίσης χρειάστηκε να παρέμβει το δούνου του και η Τρόικα. Ήταν προφανές για μας ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε στις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισαν οικογένειες και κυρίως γυναίκες. Και επικεντρωθήκαμε στο πρόβλημα του αποκλεισμού, της ανεργίας, της αύξησης των παιδιών ε, πολύ κοντά στο κατόφλι της ε, ε, φτώχειας, τα προβλήματα πιο οξυμένα για τις γυναίκες, όπου το θέμα την πρόσκαιρος συνθήκων εργασίας για τις γυναίκες εξαιτίας της πολιτικής ε, ε, που ακολουθείται για την απελευθέρωση των συνθήκων εργασία στην εργασία που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες επαναλαμβάνω η μερική απασχόληση και οι πρόσχερες συνθήκες εργασίας κατά συνέπεια αυξήθηκαν και επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από αυτά τα θέματα οι γυναίκες. Μιλούμε λοιπόν για μερική απασχόληση όταν δεν ζητείτε από τον εργαζόμενο, από την εργαζόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, το θέμα της ε, ευελιξίας στα ωράρια εργασίας, η εφαρμογή κανόνων και νόμων που αυξάνουν τα ωράρια εργασίας και τα κάνουν πιο ευέλικτα, επηρεάζει επίσης την ε, ζωή της κάθε γυναίκας και το πώς μπορεί να συνδυάσει την επαγγελματική της, την οικογενειακή και η προσωπική της ζωή μια γυναίκα. Και εδώ τίθεται θέμα ισότητας των δύο φύλων. Το 2012, τον Απρίλιο, επίσης, υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το οποίο συμφώνησαν τα δύο αυτά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν πολιτικές και προγράμματα που θα εκειώνται την ε, ε, ισότητα των δύο φύλων. Το 2012 υπεγράφει αυτό το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, αλλά δεν βλέπουμε στην πράξη να έχει εφαρμοστεί. Επίσης έχω κάνει κάποιες συμπληρωματικές ε, παρατηρήσεις που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις, την ίση αμοιβή για ίση εργασία για τα δύο φύλλα, τις αρχές για να διασφαλίσουμε τις ίση αμοιβή, να μειώσουμε την διαφορά. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ανυπαρξίας ή της μείωσης των διαθέσιμων δημοσίων υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες, η μη πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες υγείας, τα θέματα όλα που αφορούν την ε, αναπαραγωγική υγεία και την προστασία της γυναίκας. Και έθεσε στην έκθεσή μου και το θέμα της γυναίκας στην συλλογική ζωή, στην κοινωνική ζωή της κάθε κοινωνίας και στα πολιτικά. Οι γυναίκες, πρέπει να πω, ότι είναι πιο οργανωμένες. Μερικές έχουν δύο δουλειές, δεν έχουν όμως τις κατάλληλες υποστηρικτικές δημόσιες υπηρεσίες όπως ε, κέντρα φύλαξης για τα παιδιά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τρομερό πρόβλημα για τι γυναίκε που δεν μπορούν ε, έτσι να έχουν απαραίτητο χρόνο και συνθήκε να συμμετάσχουν στην κοινωνικά θέματα, στην συλλογική ζωή και κυρίω αναφέρομαι στι γυναίκε των λιγότερο ευνοούμενων στρωμάτων της κοινωνίας. Το πρόβλημα της μείωσης της ε, οικονομικής ε, δύναμης των γυναικών έχει οδηγήσει επίσης σε περισσότερες περιπτώσεις πορνείας, εκμετάλλευση των γυναικών, και έχει αυξήσει την οικονομική εξάρτηση των γυναικών που πολλές φορές εξαρτώνται πολύ περισσότερο από παλιά, από τα άτομα που τα υποχρεώνουν και τα εκβιάζουν και δεν μπορούν να ενεργήσουν ελεύθερα εναντίον τους. Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία βλέπουμε ότι όλες οι υποστηρικτικές και βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες προς γυναίκες ή ε, ΜΚΟ που είναι για γυναίκες που είναι θύματα βίας αποδυναμώθηκαν από το 2012 και μετά. Έτσι οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν είναι εξαιρετικές, κυρίως για τις γυναίκες που είναι θύματα βίας και δεν έχουν που να αποτανθούν και να επιλέξουν μια εναλλακτική στέγη σε περίπτωση βίας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα αναφέραμε, τα απαριθμίσαμε. Τα λάβαμε υπόψη και στι ανταλλαγέ απόψε που κάναμε. Και όλες οι θα έχουμε μία συνάντηση τον Ιανουάριο για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας και θα καθοριστεί βεβαίως και η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλησεν, παρακαλώ. Wasn't expecting that. Um... Α, συγγνώμη, δεν το περίμενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ζουμπέρ για το σχέδιο έκθεσης της. Ως ήθιστε βέβαια αυτό είναι ένα από τα πιο πυκνά θέματα και είναι πολύ δύσκολο να μπουν όλα στην έκθεση στο σχέδιο τουλάχιστον, οπότε πρέπει να γίνουν πολλές τροπολογίες. Α, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ. Αυτό που ελπίζω είναι να ενισχύσουμε την, ε, το αίτημα για νομοθετική δράση. Ζητάμε καθόλου τη διάρκεια αυτής της για νομοθεσία όσον αφορά την διαφορά αμοιβών, την νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, την νομοθεσία περί άδειας μητρότητας, συγγονικής άδειας. Υπάρχει επίσης ε, και το θέμα των γυναικών στα συμβούλια που έχει κολλήσει. Εντάξει, δεν έχει κολλήσει, αλλά ε, ε, με το ζόρι προχωράει, έχουμε ελπίδες. Ε, Ας ενισχυθούν λοιπόν αυτές οι πτυχές στην έκθεση. Υπάρχουν ακόμα κάποια νομικά κενά, μεγάλα. Έπειτα με εντυπωσιάζει που βλέπω πως δεν αναφέρεται πολύ το θέμα της ίσης εκπροσώπησης στην ε, λήψη πολιτικών αποφάσεων ε, εν ώψη των ε, περχόμενων εκλογών. Θα ήθελα να γίνεται μεγαλύτερη μνήμα στα πολιτικά κόμματα και έκκληση προς αυτά ώστε να φτιάξουν πιο ισορροπημένους εκλογικούς καταλόγους, μάλλον ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογέ. Να ζητήσουμε λοιπόν ισορροπημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης από άποψη φίλου. Θα καταθέσω τροπολογίες λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας άλλος τομέας που πιστεύω πρέπει να ε, αναφερθεί είναι το να συμπεριληφθεί το θέμα του φύλου στην οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να εργαζόμαστε για την κοινωνική διάσταση της ε, Νομισματικής Ένωσης, για το κοινωνικό πίνακα επιδόσεων. Επιτέλους δίνεται μια κάποια προσοχή στην κοινωνική πτυχή της οικονομικής διακυβέρνησης, οπότε τώρα ε, είναι και η ώρα να φροντίσουμε ώστε οι γυναίκες και το φύλλο γενικά, η ισότητα των φύλων να είναι ενσωματωμένα σε όλα αυτά. Γιατί όταν μιλάμε για, για ανεργία, για φτώχεια, για ανισότητα, σίγουρα το φύλλο παίζει μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά. Ε, θα καταθέσω λοιπόν κάποιες σχετικές τροπολογίες και προσβλέπω στις ε, επερχόμενες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλπάου Παραντίκα. Eh, Γεια σας, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω επιχειρήματα, αλλά πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης, εάν αφαιρέσουμε τον τίτλο και διαβάσουμε μόνο το περιεχόμενο της έκθεσης, δεν θα του βάλουμε αυτό το γενικό τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Από τη δική μας άποψη η εστίαση της εισηγήτριας γίνεται κυρίως για θέματα οικονομικά και για τις επιπτώσεις που έχουν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν αυτή τη στιγμή με την παρούσα συγκυρία μιλώ για τις γυναίκες. Τουλάχιστον όμως εγώ όταν διαβάζω τον τίτλο «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκεί που πάει ο νους μου είναι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για μία πρωτοβουλία συνολική στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία δομή που να ε, εφαρμοστεί υποχρεωτικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνειδητοποιώ βεβαίως ότι πρέπει να είναι σύντομο το κείμενο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για μία δομή νόμου, της Ευρω... Ε, μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μου λείπει λοιπόν εμένα. Δεδομένου ότι υπάρχει σαφής ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση ισότητος. Για τον ε, παιδεία, για την κατάρτιση δεν αναφέρουμε τίποτα. Για την ε, γλώσσα που χρησιμοποιείται στην σεξιστική πολλές φορές. Ε, και να αναφέρουμε τουλάχιστον ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τέτοιες σεξιστικές εκφράσεις, τέτοιο λεξιλόγιο. Πολλές φορές ε, παραφανίζεται αυτό σαν καρικατούρα, αλλά ώρες ώρες είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σοβαρά, όπως είχαμε εμείς ε, προβλήματα στην βασική χώρα. Ο πρόεδρος Ιμπαρέτσε αποφάσισε να λέει ή, οι άντρες και οι γυναίκες ε, και σήμερα ακόμη και Καρικατούρα έγινε αυτό και αστείο. Και σήμερα η... στην ε, βασκική χώρα δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Άρα η παιδεία, η ανάγκη να υπάρχουν συντονισμένα μέτρα, η χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου, η παροχή υπηρεσιών, η φροντίδα των παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων, ο καθορισμός κάποιων ε, ε, και ωραρίων ώστε να μπορούν να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους οι γυναίκες. Η συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα ώστε σε κάθε χώρα να υπάρχουν νόμοι που να επιτρέπουν το περίφημο πρόβλημα της ποσόστοσης να είναι πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε μόνο αρνητικά την παρουσία των γυναικών, αλλά και τα θετικά. Τι έχει γίνει. Πολλές φορές με το θετικό κάνουμε κάτι καλύτερο, Πώς είναι παρούσες ακόμη και σε διοικητικά συμβούλια γυναίκες, να τονίσουμε αυτή την διάσταση θετική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις για το τι ακριβώς θα θέλαμε να γίνει συσφαιρικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε χώρα. Γι' αυτό, για μένα, η ανισότητα ε, οδηγεί στα αποτελέσματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση, οδηγεί σε κακομεταχείριση, αλλά θα πρέπει να πούμε και ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υιοθετηθούν σε κάποιες χώρες, διότι υπάρχουν ε, χώρες που δεν έχουν ακόμη ε, μέτρα προστασίας για τις γυναίκες σε τέτοιες περιπτώσεις βίας. Και γιατί να μην μιλήσουμε και για μία νέα πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να σταματήσουμε να ε, χρησιμοποιούμε τα στερεότυπα που χρησιμοποιούν ακόμη και κάποιες ενώσεις τις οποίες, ε, ή κάποιοι όμιλοι στους οποίους υπάρχουν μόνο άνδρες, μόνον άνδρες και λένε ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγανε στο παρελθόν. Και μιλούμε για δύο φύλλα, αλλά μιλούμε για κάτι πολύ πιο ευρύ σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση και εστίαση στην έκθεση αυτή, ώστε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα μας οδηγήσει να κάνουμε κάτι από κοινού για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της ανισότητας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ κυρία Αντίτα Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και να πω ότι θεωρώ ότι το τμήμα των προτάσεων είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το τμήμα της διάγνωσης της κατάστασης. Αυτή η διαδικασία που εμείς ε, παρακολουθούμε και την πρόθεση δηλαδή των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα γίνεται από ε, βήματα μπροστά αλλά και βήματα πίσω κάποιες φορές ε, και νομίζω πως σχετικά σε σύγκριση με το 2000 2009-2007 θα έτεινα να συμπεράνω ότι υπήρξαν περισσότερες ε, οπισθοδρομήσεις παρά πρόοδοι. Υπήρξαν κάποια καλά παραδείγματα κάποιων νομοθεσιών που καταρτίστηκαν, αλλά υπάρχουν ωστόσο και παραδείγματα νομοθεσίας που θα ήθελα να είχαν εγκριθεί αλλά που δυστυχώς μπλοκαρίστηκαν στο Συμβούλιο. Οδηγίες όπως η άδεια μητρότητας. Πιστεύω μάλιστα πως γενικά σε αυτό το τομέα υπήρξε λιγότερες φιλοδοξίες και λιγότερες πρόοδοι από ό,τι στο παρελθόν. Και μπορούμε να το παρατηρήσουμε αυτό και στην ε, επιμονή των στερεοτύπων ε, λόγω φύλου. Για παράδειγμα, αν δει κανείς διαφημίσεις, ε, το διαπιστώνει αυτό, αλλά και στο επίπεδο της παιδείας, στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως αυτή αναμεταδίδεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια και οι ανισότητες οι οποίες επικρατούν συνδέονται πάρα πολύ στενά με την οικονομική κατάσταση, αύξηση της βίας. Υπάρχουν μελέτες πρόσφατες που αποκαλύπτουν ότι υπήρξε αύξηση της ε, κατοίκων βίας, πράγμα που σχετί... όχι μόνο απέναντι στις γυναίκες αλλά και στα παιδιά απέναντι. Και υπήρξε αύξηση της ανισότητας στην υγεία, δηλαδή οι γυναίκες έχουν ακόμη περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγείας, ε, κυρίως υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και άλλη μια πτυχή που αποκαλύπτεται από τη μελέτη και που έγινε πρόσφατα και είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ ανησυχητικό, είναι αυτό που αφορά το ποσοστό γεννητικότητας. Δηλαδή, σε αυτή τη μελέτη αναφέρεται ότι οι γυναίκες τα ήθελαν να έχουν περισσότερα παιδιά, αλλά ότι δεν μπορούν, για να, δεν μπορούν. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση, κατά τη γνώμη μου γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν οι συνθήκες, να πληρούνται οι όροι, ώστε οι οικογένειες και οι ευρωπαίες γυναίκες που θέλουν να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για άλλους δείκτες που αποκαλύπτουν δυστυχώς ότι δεν προοδεύουν τα πράγματα. Και εμείς εδώ στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέπουμε ότι υπάρχει λιγότερη προσοχή και λιγότερη ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα. Ε, οι πολιτικές, οι κοινωνικές δυστυχώς ε, κυριαρχήθηκαν από άλλα θέματα και έπεσαν σε δεύτερο πλάνο. Η ευρωπαϊκή ατζέντα είναι γεμάτη με τα οικονομικά θέματα. Άντε και λίγο περιβάλλον αλλά τα κοινωνικά θέματα έχουν μπει σε δευτερεύοντα ρόλο. Και μέσα στα κοινωνικά θέματα η ισότητα των φίλων έχει και αυτή ο ε, οπισθοχωρήσει ως θέμα, δεν είναι πια θέμα προτεραιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον από την Κομισιόν εδώ που να θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Δεν είναι κανείς εδώ. Α, παρακαλώ. Ε, σας έψαχνα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να πάρουμε το λόγο για το θέμα της ισότητας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες το 2012. Η Κομισιόν δημοσίευσε την ετήσια έκθεση τον Μάιο του 2013 για την κατάσταση του 2012. Η έκθεση αυτή είναι βασισμένη στις προτεραιότητες και τις στρατηγικές για την ισότητα γυναικών ανδρών, τονίζοντας τα σημεία που θεωρήσαμε ότι ήταν τα πιο σημαντικά. Το πιο... Ένα από αυτά ήταν η επίπτωση της οικονομικής κρίσης ε, στην ισότητα, βλέπουμε πως οι ανισότητες ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες έχουν ε, υποχωρήσει στο οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ε, αλλά αυτό δεν οφείλεται στην βελτίωση της κατάστασης της γυναίκας, αλλά στην ταχύτερη επιδείνωση της κατάστασης των ανδρών. με άλλα λόγια, βλέπουμε μια εξίσωση προς τα κάτω όσον αφορά την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της απασχόλησης, των μισθών, των αποδοχών και της στόχιας και οι ε, αποστάσεις είναι σημαντικές 12% όσον αφορά την απασχόληση 16% όσον αφορά τις αποδοχές και πάλι λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε τις πιο ευάλωτες ομάδες δηλαδή τους νέους που πλήττονται από την κρίση και γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες είναι πιο ε, πιθανόν να βρεθούν εκτός της αγοράς εργασίας Δηλαδή δεν μπορούν να βρουν ούτε δουλειά ούτε κάποια μαθητεία είτε κατάρτιση και είναι και λιγότερες ε, που λαμβάνουν ε, στήριξη δημόσια, δηλαδή ε, κάποια κατάρτιση ή μαθητεία ή βοήθεια. Οι ανισότητες αυξάνονται λοιπόν και με την γέννηση παιδιών και τονίζονται καθώς προχωράει η ζωή και για πρώτη φορά δημοσιεύσαμε έναν αριθμό ε, όσον αφορά τη διαφορά στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών που φτάνουν στο 39%. Πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή. Τα μέτρα που υπάρχουν για την ενίσχυση της ε, ισότητας ανάμεσα στις άντρες και την των ανδρών υπάρχουν πολλά μέσα, δηλαδή διεύρυνση των μέσων φροντίδας για τα παιδιά και η απασχόληση να, είναι, να δίνει τις ίδιες αποδοχές σε άνδρες και γυναίκες για ίση εργασία και αυτές οι συστάσεις έχουν ε, προταθεί στις χώρες μέσα στο πλαίσιο του εξαμήνου, του, 12, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2012 και το 2013 εκ νέου υποβλήθηκαν αυτές οι προτάσεις. Ξέρουμε ότι πρέπει να συνδυαστεί το ευρωπαϊκό επίπεδο με το εθνικό για να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών. Υπάρχουν πολύ καλές πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο παρατηρούμε ότι τα καταφύγια για τις γυναίκες και τα οι αριθμοί, τηλεφωνικοί αριθμοί επίγουσας ανάγκης που είναι τα πιο κοινά μέσα για την καταπολέμηση της βίας δεν υπάρχουν παντού. Δηλαδή πρόκειται για μια ανέκθεση που έδειχνε ε, τις που έχουν επιτευχθεί αλλά και τις πρόοδες που πρέπει ακόμα να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σούπερ για να κλείσει. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω και όπως είπε και η πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η έκθεση αυτή γίνεται με βάση την αξιολόγηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισότητα των δύο φύλων το 2012. Δηλαδή, ακολουθείται η δομή της έκθεσης της Κομισιό με μικροδιαφορές και πολλά ε, σχόλια έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση αυτής της διάγνωσης που είχε γίνει τότε. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι συνεισφορές των συναδέλφων ήταν θετικές και σημαντικές. Αυτό το λέγω όμως για να εξηγήσω λίγο τα πλαίσια μέσα στα οποία ε, συντάχθηκε η έκθεση αυτή. Και όπως σας είπα επίσης, και είναι και θέμα σύνταξης. Δεν, μπορώ να συμπεριλάβω, δεν μπορούσα να συμπεριλάβω τα πάντα. Θα είναι πολύ πιο τελειοποιημένη στο τέλος η έκθεση. Αλλά επειδή η έκθεση της Επιτροπής βασίστηκε στα οικονομικά κριτήρια και επιπτώσεις και εγώ το έκανα γιατί είναι και επίκαιρο θέμα σήμερα. Ίσως η δική μου η προσέγγιση εξαρτάται και από την πραγματικότητα στην οποία ζω. Και όλοι μας θα υποφέρουμε από αυτό το πρόβλημα, διότι οι ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλές μεταξύ κρατών, εντός των κρατών κτλ. Όλους λοιπόν μας επηρεάζει αυτό το θέμα κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ το οποίο είναι και αμφιλεγόμενο. Όπως έλεγε η Εντίδε Στρέλα. Πριν από μερικά χρόνια μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα. Για διαφορετική συμπεριφορά, για στερεότυπα. Σήμερα όμως οπισθοδρομήσαμε Και για πολλές γυναίκες οι βασικές διεκδικήσεις ακόμη τίθενται ένα αμφιβόλο. Σήμερα λοιπόν έτσι ζούμε αυτή την κατάσταση και δεν νομίζω ότι μπορούμε να μην το τονίσουμε αυτό. Βεβαίως είμαι στην ε, διάθεση όλων και περιμένω να κατατεθούν από τις συναδέλφους οι τροπολογίες για να τις συμπεριλάβω στην εκθεσία μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 18 Δεκεμβρίου στις 12 και θα συζητήσουμε τις τροπολογίες 22-23 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε επίσης 22-23 Ιανουαρίου. Στην Ολομέλεια θα πάει τον Μάρτιο. Ολοκληρώσαμε στο σημείο 6 και περνάμε στο σημείο 7. Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην ισότητα των φίλων Και δίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Χάνιμπολ. Εκτός μικροφώνου. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση αυτή εδώ σε σας. Χαίρομαι που η Γαλλική Διεθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νόμο όπου υιοθετεί το σουηδικό μοντέλο πριν λίγες μέρες. Υπάρχει λοιπόν όχι μόνο ενδιαφέρον αλλά και επιθυμία να ε, καταπολεμηθεί η πορνεία και η ανισότητα και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη η έκθεση αυτή και ελπίζω να την ε, υπερψηφίσετε. Η έκθεση αυτή βασίζεται στο ότι η πορνεία είναι ένα, μια ε, έκφανση της ανισότητας των φύλων και αν είχαμε ισότητα δεν θα είχαμε και πορνεία. Διότι οι άνδρες αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες από τις γυναίκες και μπορεί κάποιος να σας πει ότι μερικές φορές ε, συμβαίνει το αντίθετο, αλλά μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσεις. Είναι λοιπόν ε, θέμα ανισότητας μεταξύ των φύλων και θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Να μιλάμε για την πορνεία ως μορφή βίασης βάρος των γυναικών, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών ε, που εκπορνεύονται δεν θέλουν ε, να το κάνουν. Κατά τη διάρκεια ε, σύνταξης αυτής της έκθεσης είχα διάφορες συναντήσεις με όσους συμμετέχουν σε αυτά, με όσους ασχολούνται με αυτά και Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που υποστηρίζουν ότι ε, εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ, όπως την ονομάζουν, ε, από επιλογή, αλλά είναι πολύ μικρή μειονότητα. Υπάρχουν πολλοί που αναγκάστηκαν ε, να καταλήξουν εκεί, υπάρχουν κάποιοι που λόγω φτώχειας δεν είχαν άλλη επιλογή και μεγάλο ποσοστό ε, των γυναικών παίρνουν και ναρκωτικά διότι είναι τόσο άσχημη η κατάσταση, είναι τόσο ελεηνές οι συνθήκες που χρειάζεται κάπως να ξεφύγουν. Είναι κάτι λοιπόν που επηρεάζει όλο τον κόσμο, αλλά επηρεάζει ιδιαίτερα τις μεγάλες ε, πόλεις της Ευρώπης. Και φυσικά υπάρχει κάποια σχέση με την εμπορία ανθρώπων, κάτι που πάντα με απασχολούσε, διότι πολλές γυναίκες θύματα της ε, Εμπορία ανθρώπων ε, προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη και καταλήγουν ε, στο Λονδίνο. Το έχω δει αυτό με τα ίδια μου τα μάτια. Το 76% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό ε, δείχνει ακριβώς ότι η πορνεία είναι είδος βίας. Πρέπει όμως να θέσω και το αντεπιχείρημα. Υπάρχουν δύο θεωρίες ή δύο θέσεις που αφορούν την πορνεία. Η μία, την οποία υποστηρίζω εγώ, είναι ότι η πορνεία είναι καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ελαχιστοποιήσουμε την πορνεία. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη οπτική διαφορετικό μοντέλο που υποστηρίζει ότι η πορνεία υποστηρίζει την ισότητα των φύλων, διότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να ε, επιλέξουν τι θα κάνουν με το σώμα τους. Ε, και αν το επιλέγουν θα πρέπει ε, να τους επιτρέπουμε την επιλογή αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση και προτού προχωρήσουμε περισσότερο, αξίζει τον κόπο να κοιτάξουμε τον νόμο περί πορνείας στα διάφορα κράτη-μέλη. Περισσότερα γνωρίζω προφανώς ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου επικρατεί μεγάλη σύγχυση στον νόμο. Η πορνή αυτή καθεαυτή δεν είναι νόμιμη. Θεωρείται έγκλημα, όλα όμως όσα σχετίζονται με αυτήν είναι νόμιμα. Οπότε η Και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες είναι τα θύματα και αυτό είναι το θέμα παντού όπου είναι παράνομη η πορνεία, ότι οι γυναίκες καταλήγουν να είναι τα θύματα. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Ιρλανδία. Παρ' όλα αυτά εξετάζεται εκεί η δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης, αλλαγής της κατάστασης. Η Γαλλία έλαβε αυτήν την σημαντική απόφαση. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι νόμιμη η πορνεία οι χώρες για τις οποίες ακούμε περισσότερα είναι οι κάτω χώρες και η Γερμανία. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι δύο αυτές χώρες νομιμοποίησαν αρχές του 2000 ε, την πορνεία, αλλά έχουν αρχίσει να το μετανιώνουν. Οι κάτω χώρες έχουν γίνει ο κατεξοχήν προορισμός για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Έχουν περίπου 7.000 άτομα το χρόνο και έχω ακούσει ε, παρατηρήσεις ε, του Δημάρχου του Άμστερνταμ που έχει καταλήξει η σεξουαλική πρωτεύουσα της Ευρώπης ε, και δεν του αρέσει η κατάσταση. Στην Γερμανία υπάρχουν 400.000 πόρνες, 20, 20 φορές περισσότερο από ό,τι στη Γαλλία, ακόμα και πριν αλλάξει η Γαλλία τον σχετικό νόμο. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η νομιμοποίηση της πορνείας δεν έχει βοηθήσει. Αντιθέτως, έχει επιδονώσει την κατάσταση. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια όταν ε, οργανώθηκε το παγκόσμιο κύπελο στο Μόναχο, υπήρχαν αιτήματα από τον κόσμο, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί οίκοι και αύξηση της πορνείας, επειδή ακριβώς υπήρχαν περισσότεροι πελάτες. Δεν θα ήθελα να φαίνεται σαν να μας συγχαίρω. Επειδή η πορνεία όμως δεν είναι νόμιμη ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, στο Λονδίνο με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών δεν είχαμε παρόμοια προβλήματα. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να καταλήξουμε κάπου να έχουμε ένα πρότυπο αντιμετώπισης της πορνείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρ του μοντέλου που έχει οθετήσει η Σουηδία και που αν περάσει από τη Γερουσία θα ε, περάσει και στη Γαλλία και που ε, ε, έχει χρησιμοποιήσει και η Νορβηγία και η Ισλανδία που ουσιαστικά καθιστά εγκληματίε όσους αγοράζουν τέτοιε υπηρεσίες, του άντρε, δηλαδή. Έτσι, ο πελάτης δεν πρέπει να το κάνει, το οποίο ακριβώς σημαίνει ότι δεν γίνονται θύματα οι γυναίκε. Και από την θέση σε ισχύ του νόμου στη Σουηδία είδαμε μεγάλη πτώση στον αριθμό των γυναικών που εκπορνεύονται στους δρόμους. Και αυτό θέλουμε να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι η πορνεία αντίκειται στην ισότητα των φύλων και ως Επιτροπή Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να μειωθεί η πορνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή. Δίνω τώρα το λόγο. Ε, πρώτον, στην κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιάδης η η κυρία Λούνατσεκ είναι, αλλά δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα και την αντικαθιστώ. Δεν είναι μυστικό ότι εγώ ήμουνα τη άποψη ότι έπρεπε να γίνει αυτή η έκθεση, κυρίω αυτή την εποχή προεκλογικής εξαρτία, διότι θα δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ των διαφόρων ομάδων με αντιμαχόμενες ιδέες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα εθνικό του καθένα. Οι Γάλλοι πάνε προς μια κατεύθυνση, η δική μου η χώρα, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί διαλέγουν κι άλλη, άλλη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, τελικά δεν νομίζω ότι τελικά θα πρόκειται για κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στην προεκλογική μας εκστρατεία πολύ. Αλλά είμαι όπως λέει το. Δεν είμαι όπως το ε, ΕΛΚ στην ε, περίπτωση των ε, LGBT και αυτή την πολιτική που ακολούθησαν. Έχουμε ανοιχτό πνεύμα για αυτό το θέμα. Ε, έχουμε εδώ να κάνουμε με την καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι το βλέπουν οι Γάλλοι, οι Σουηδοί το βλέπουν διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ότι ε, πρέπει να το δούμε από την μεριά των γυναικών. Η δική μου η μητέρα ξέρω ότι αγωνίστηκε για να είναι αυτή που αποφασίζει για το τι θα κάνει το σώμα της και έτσι πρέπει να είναι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις που είναι δυνατές ανοιχτές. Βεβαίως συμφωνούμε μεταξύ μας ότι οποιαδήποτε μορφή υποχρεωτικής πορνείας και εμπορίας ανθρωπίνων όντων ε, θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Αυτού του είδους η πορνεία θα πρέπει να καταπονηθεί και αν πρόκειται να κάνουμε ε, κάτι γενικότερη την πορνεία ίσως και μόνο θα μπορούσα να συμφωνήσουμε σε περισσότερα θέματα. Τέλος πάντων δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα μπορούσα να το κάνω αλλά ως τελευταία παρατήρηση επιτρέψτε μου να πω ότι όντως συμφωνούμε ότι ίσως πολλές γυναίκες που εργάζονται στον τομέα της πορνείας θα προτιμούσαν να κάνουν μια άλλη δουλειά. Αν τους απέφερε η άλλη δουλειά τόσα πολλά χρήματα θα τους αποφέρει αυτή τους η δραστηριότητα. Ας είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να δώσουμε αυτή την επιλογή στις γυναίκες. Με καλύτερη μόρφωση, με προγράμματα που μπορούν να τις αποσπάσουν από την πορνεία αν το θέλουν, με δημιουργίες νέων θέσεων απασχόληση. Αντί λοιπόν να κλείνουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και να τις οδηγούμε στην φτώχεια, ας κάνουμε κάτι το πιο θετικό. Ας προσπαθήσουμε. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα σημεία στα οποία συμφωνούμε και νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πολύ εάν σε πολλά σημεία της έκθεσης μιλούσαμε για ε, αναγκαστική πορνεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Οβίρ. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση της ε, στην έκθεση της ηγήτριας είναι σωστή, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης προς την ε, πορνεία ως εμπόδιο για την προώθηση της ισότητας. Σχεδόν το 95% των ε, εκδιδόμενων γυναικών έχουν υποφέρει από κάποιο είδος βίας στο παρελθόν. Οι περισσότερες πόνες προέρχονται από χώρες όπου επικρατούν πολύ χαμηλές ε, προδιαγραφές διαβίωσης και γι' αυτό στην ουσία είναι οικονομικοί όμοιροι, είναι θύματα ούτως ή άλλως. Το 90% εξ αυτών εξαρτώνται από ε, από μαστροπούς που τις χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Ε, και σε μεγάλο βαθμό η πορνεία ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα και περιλαμβάνει ψυχική και σωματική βία. Ε, αυτά όλα είναι καθημερινά σε την περίπτωση, σε, την, σε αυτόν τον κλάδο. Οι αντιδράσεις μας μπορεί να είναι εξή. Καταρχήν, να νομιμοποιηθεί τόσο η πορνεία όσο και η μαστροπία. Δεύτερον, να ε, ποινικοποιηθεί μόνο η μαστροπία. Τρίτον, χώρες όπου το, η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είναι ε, ποινικοποιημένη, η πορνεία να είναι αποποινικοποιημένη. Βλέπουμε ότι στα κάτι μέλη της πρώτης ομάδας υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες ενδείξεις ότι αυτή η στάση δεν είναι βάσιμη. Στη δεύτερη ε, περίπτωση, εκεί όπου έχει ποινικοποιηθεί η μαστροπία, ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Για παράδειγμα, στη δική μου χώρα, την Εστονία, οι πόρνες τώρα καταγράφονται ως αυτοαπασχολούμενες, αλλά οι μαστροποί παραμένουν και τις ελέγχουν πίσω από την πλάτη τους, σαν σκιές. Όμως η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι αποτελεσματική. Γι' αυτό πιστεύουμε πως μόνο η ποινικοποίηση της αγοράς ε, σεξουαλικών υπηρεσιών και της μαστροπίας μπορούν να λειτουργήσουν. Με, στη γλώσσα της οικονομίας της αγοράς, εάν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει και παροχή. Ως ρεαλίστρια γνωρίζω πως αυτό δεν θα είναι εύκολο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε κάθε πολιτική ομάδα συμπεριλαμβανομένες της ΑΛΔΕ. Και σίγουρα θα υποβάλουμε και εμείς κάποιες προτάσεις για τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για την Σκανδιναβία, για την κυρία Κορνέλισεν. Στην Δανία δεν είναι παρανομή η πορνεία. Στη Δανία απαγορεύεται η μαστροπία, αλλά το ε, να είναι κανείς πόρνη είναι ε, νόμιμο. Και επίσης το να έχει κανείς οίκο είναι ε, παράνομο, ε, δηλαδή το να βγάζει κανείς ε, χρήματα επειδή εκπονεύεται κάποιος άλλος είναι παράνομος. Και επίσης η, φορολογία θέλει η εφορία θέλει πολύ τα φορολογικά έσοδα από την πορνεία. Είμαστε λοιπόν μεγάλη πλειοψηφία στο Δανέζικο Κοινοβούλιο είναι κατά του να είναι παράνομη η πορνεία. Νομίζω ότι η νομιμοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το να θεωρείται μια κανονική δουλειά. Δεν μπορεί όμως να πάει κανείς σε γραφείο της εργασίας και να ε, του του προτείνουν μια τέτοια δουλειά και επίση θα πρέπει να είναι ασφαλή κανεί στον χώρο εργασία του. Στην προηγούμενη θητεία, μια συναδελφο από την ομάδα S&D ήταν, από την Αυστρία ήταν υπέρ τη ελεύθερη πορνείας και ε, συνέταξε μια έκθεση για την βία εις βάρος ε, των γυναικών που εκπορνεύονται. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Δανία έφτιαξε μια ταινία για τρεις πόρνες και ήταν και οι τρεις υπέρ. Μία από αυτές είπε είμαι πάρα πολύ απασχολημένη, έχω τέσσερα παιδιά και είναι δύσκολη η δουλειά. Κάθε μέρα με βιάζουν, κάθε μέρα με δέρνουν, με έχουν ταγκώσει και κοντέψαν να με πνίξουν, να με απαγχωνίσουν. Να, να Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε την πορνεία με μια κανονική δουλειά. Εάν στο κέντρο εξέβρεση εργασία ε, μπορεί κανεί ε, να κάνει αίτηση για μια τέτοια δουλειά, τότε είναι μια δουλειά όπω όλε οι άλλε. Αλλά ο κόσμο είναι υποκριτέ. Χρησιμοποιούν διπλά μέτρα και σταθμά. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις στατιστικές. Η γαλλική κυβέρνηση λέει ότι το 90% των γυναικών που εκπονεύονται στη Γαλλία είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η Βρετανική αστυνομία λέει ότι το 80% είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή έχουν μαστροπό. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρούμε αυτήν την ελεύθερη άσκηση του επαγγελματο και η Γαλλία υιοθέτησε την νομοθεσία αυτή λόγω Τη εμπορία ανθρώπων. Βρέθηκα στη Ρουμανία και συνομίλησα με πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις που φροντίζουν τι γυναίκε θύματα εμπορία ανθρώπων και μας λένε ότι ο αριθμός των γυναικών αυτών στις χώρες όπου είναι νόμιμη η πορνεία είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλες χώρες. Η εμπορία ανθρώπων είναι σημαντικό πρόβλημα και στις κατοχώρες και στην Γερμανία όπου είναι νόμιμη η πορνεία. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και αυτό. Και τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει η υποκρισία. Εάν θέλουν ελεύθερη πορνεία, εάν θέλουν να θεωρείται κανονική δουλειά, εντάξει, αλλά τότε θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χειρίζονται και τα κέντρα ευρέσεως εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο από την Κομισιόν, η κυρία Φαστρέ, παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Η κυρία Σούπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εμείς ε, είμαστε υπέρ της εξής προσέγγισης. Πρέπει η μαστροπία να ποινικοποιείται και να ποινικοποιείται το άτομο το οποίο οδηγεί στην πορνεία. Είναι θύμα ο άνδρας ή η γυναίκα που οδηγείται στην πορνεία. Και είναι θέμα βίας. βία δεν μπορεί να είναι οικειοθελής ή εξαναγκαστική. Η εργασία δεν είναι μόνο, δεν έχει ως μόνο στόχο να κερδίσει κάποιος χρήματα. Είναι ένας τρόπος για να ολοκληρωθεί κανείς ως άτομο και δεν νομίζω ότι κάποιος είναι, κάποια γυναίκα είναι παραγωγική και ανθίζει ως προσωπικότητα όταν ένας άνδρας αγοράζει τις υπηρεσίες της. Συμφωνούμε λοιπόν. Γενικά, ίσως όχι με όλα όσα λέγονται, δεν θα χρησιμοποιήσω επιχειρήματα που βασίζονται σε στατιστικές, αλλά διαβάζοντας την έκθεση μου ήρθαν κάποιες ιδέες για την κατάθεση τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε νέα φαινόμενα που εμφανίστηκαν πάρα πολύ πρόσφατα σε σχέση με την πορνεία και κυρίως φαινόμενα σύμφωνα με τα οποία διάφορες γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικονομικά στρώματα ε, ε, εκδίδονται εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων των σημερινών. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διασυνδέσουμε το θέμα αυτό με την κοινωνική συμπερίληψη με την εκπαίδευση, με συνοδευτικά μέτρα εκ μέρους των κρατών, όχι μόνο για να προβλεφθεί μια άλλη πηγή εισοδήματος για τέτοιου είδους γυναίκες, αλλά και άλλα συνοδευτικά μέτρα για να βοηθηθούν. Επίσης, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι ενώσεις και οι οργανώσεις ε, οι οποίες ε, φιλοξενούν γυναίκες που έχουν ε, ε, εργαστεί ως πόρνες, αλλά καταλήγουν σε αυτές τις οργανώσεις για να προσφεύγουν σε αυτές τις οργανώσεις για να προστατευτούν. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μικρές αγγελίες πώληση τέτοιου είδους υπηρεσιών εντός εισαγωγικών που το διαβάζουμε στις κανονικές εφημερίδες πλέον και στα περιοδικά σήμερα ξέρω τι ισχύει για την κάθε νομοθεσία, αλλά στη χώρα μου, σε οποιαδήποτε πλέον εφημερίδα ή εβδομαδιαίο περιοδικό, διαβάζουμε σε μία σελίδα κάτι για την πρόσφυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην επόμενη σελίδα έχουμε φωτογραφίες σεξι διαφόρων γυναικών που πολλούν τις υπηρεσίες τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να θέσουμε για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν, την κυρία Φραστρέ, παρακαλώ. Thank you very much for giving... Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat του Απριλίου 2013, η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εμπορίας ανθρωπίνων όντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα, ε, η πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία φορά τις γυναίκες, σε ποσοστό 96%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την πάση σχέση μεταξύ εμπορίας μεταξύ γυναικών και πορνείας. Όσον αφορά τις πολιτικές, δηλαδή της πορνείας, αυτές είναι θέμα αρμοδιότητας κάθε κράτους μέλους χωριστά και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι εθνικές προσεγγίσεις για τα θέματα πορνείας, η εθνική νομοθεσία και η πρακτική τους εφαρμογή διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη η... Ακόμη και η πρακτική εφαρμογή των νόμων, ακόμη και εντός των ίδιων των χωρών, μπορεί πολλές φορές να είναι αντιφατική. Αυτές οι εθνικές προσεγγίσεις διαμορφώνονται από τις ε, παραδόσεις, τις ε, πολιτικές και τις διάφορες ε, θεωρήσεις και τις συνήθειες κάθε χώρας. Τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε με εμπορία ανθρωπίνων όντων, έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει ένα ε, πλαίσιο νομοθετικό για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου με τη σχετική οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας των ε, ανθρωπίνων όντων, όπου το κέντρο εδώ είναι το ανθρώπινο ε, θύμα. Um, και θα ήθελα να σας πω ότι έχουν εμπεριστατωμένες νομοδοτήσεις σταλεί σε χώρες οι οποίες δεν έχουν προβλέψει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα πώς διαμορφώνεται και η ζήτηση. Η οδηγία δημιουργεί την ε, ε, νομική υποχρέωση των κρατών μελών να μειώσει τη ζήτηση. Και ζητεί η οδηγία επίσης τα κράτη-μέλη να το θεωρήσουν αυτό ως ένα ε, ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με την οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αναφορά επί αυτού του θέματος της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από μερικά χρόνια για τα μέτρα που προβλέπονται και δέχτηκε προτάσεις για κάθε γυναίκα που ασκεί αυτό το επάγγελμα υπάρχει κάποιος ο οποίος ζητά τις υπηρεσίες της. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα και δύσκολα θέματα όπως Φερρυπίν σε ποιο άλλο τομέα της εγκληματικότητας δεν ποινικοποιείται αυτό το αδίκημα. Στα πλαίσια της τριγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, κρίζωση ε, της εμπορίας ανθρωπίνων όντων 2012 και 2016 προβλέπονται μέτρα τα οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εξειδικευμένοι οργανισμοί και τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια στρατηγική που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο του 2012. Πολλές από τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν σε αυτή τη στρατηγική έχουν σχέση με την σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών, όπως η πρόληψη, οι έρευνες ε, ανάλογα με τα δύο φύλλα, η σωστή κατάρτιση κτλ. Επίσης, στην στρατηγική αυτή εντοπίζονται και δράσεις ώστε με κάποιες επιμένες τρίτες χώρες να μπορέσουμε να λύσουμε καλύτερα το πρόβλημα της πορνείας. Επίσης, η μελέτη σχετική με την εμπορία ανθρωπίνων όντων, που όταν θα έχει ολοκληρωθεί, θα δούμε περισσότερο πώς συνδέεται αυτό το θέμα με την εκμετάλλευση των δύο φύλων και το πόσο ευάλωτες είναι και ευάλωτα είναι τα άτομα τα οποία είναι θύματα πορνείας. was μια δεύτερη εφαρμοστική έκθεση εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και συμπεριλαμβάνονται περιοχές και χώρες κατά προτεραιότητες με τις οποίες θα πρέπει να ενταθεί η συνεργασία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της εκμετάλλευσης ανθρωπίνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μπορέσουν να κάνουν μία χαρτογράφηση της όλης κατάστασης και να μπορέσουν να δούνε πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν εδώ και τα κράτη-μέλη και πώς θα μπορέσει να γίνει και συνεργασία με τρίτες χώρες και περιοχές για να μπορέσουμε τις δεσμεύσεις να αναλάβουμε να τις κάνουμε συγκεκριμένες και λειτουργικές. Επιτρέψτε μου επίσης να πω και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται τα θύματα και στα πλαίσια του προγράμματος Δάφνη, η Επιτροπή χρηματοδότησε μία σειρά σχεδίων με στόχο την γυναικεία πορνεία, δεδομένου ότι πρόκειται για μία ομάδα ευάλωτη και εκτεθειμένη στη βία. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω την ε, θέση του συντονιστή τη Ευρωπαϊκή για τέτοιου είδους θέματα. Είναι κάτι το οποίο προβλεπόταν καταρχάς στο πρόγραμμα τη ΟΧΟΛΜΗΣ και μετά εκπονήθηκε ε, και οριστικοποιήθηκε στα πλαίσια της σχετικής οδηγίας του 2012 θα είναι υπεύθυνο ή υπεύθυνη για την βελτίωση του συντονισμού και της συνεκτικότητας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών και των διεθνών φορέων και θα έχουμε μια νέα πολιτική στον τομέα αυτό. Ως η συντονιστής είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και εφαρμόζει τη νέα ε, ενοποιημένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίδει τους γενικούς προσανατολισμούς για την ε, εκτός συνόρων ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτική. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι προσπαθώντας να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, ίσως θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε περισσότερο στις κοινέ προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για να εκριζωθεί αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ. Thank you so much for that. And σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ πολύτιμες πληροφορίες μας δώσατε και σχετικά με την θέση της Κομισιόν. Προσωπικά, με ενδιαφέρον τα επιχειρήματά σας για τη ζήτηση που αποτελεί σημαντικό μέρος της συζήτησης όταν μιλάμε για την πορνεία. Τονίσατε όμως και τη σχέση ανάμεσα στην πορνεία και την εμπορία ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στην κυρία Χάνιμπολ για να κλείσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν. Ήταν πολύ ε, χρήσιμα αυτά που μας είπε και έθεσαν την όλη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για την ισότητα, αλλά μιλάμε και για την εμπορία ανθρώπων. Αναφέρατε τα στοιχεία το, της Κομισιόν. Το 96% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ε, θύματα απορνίας και Σε μία από τις προηγούμενες παρεμβάσεις ακούσαμε για την διαφήμιση των σεξουαλικών υπηρεσιών σε εφημερίδες. Περίπου πριν τρία χρόνια έκανα σχετική έρευνα. Η αστυνομία στο Λονδίνο είναι απολύτως πεπισμένη ότι υπάρχει άμεση σχέση και ότι αυτές οι διαφημίσεις διαφημίζουν υπηρεσίες από γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Όλο αυτό το επιχείρημα λοιπόν που αφορά την εμπορία ανθρώπων είναι ο βασικός λόγος που θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Και έχει να κάνει και με την καταναγκαστική πορνεία, διότι εάν το 96% των γυναικών αυτών είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, τότε προφανώς είναι θύματα καταναγκασμού. Οι γυναίκες αναγκάζονται παρά τη θέλησή τους να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Και πολύ μικρός αριθμός επιλέγει πραγματικά να το κάνει και θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό ούτως ή άλλως. Δεν θέλει κανείς να τη σταματήσει και η πλευρά της ζήτησης είναι επίση σημαντική. Εάν δεν υπάρχει ζήτηση θα, πέσει και, θα μειωθεί και η εμπορία ανθρώπων. Υπάρχουν ε, στοιχεία που δείχνουν ότι το μοντέλο της Σουηδίας, το σουηδικό πρότυπο, έχει μειώσει τη ζήτηση. Καταλαβαίνω ότι το θέμα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι όμω επίση σαφέ ότι υπάρχει αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη διασυνοριακή φύση και τη εμπορία ανθρώπων. Θα ήθελα να πω κάτι στο οποίο έπεσε την προσοχή μα η Μπρίτα Τόμσον. Η πορνεία δεν είναι μια κανονική δουλειά. Δεν πηγαίνει κανεί σε γραφείο εξεύρεση εργασία και λέει ότι εγώ αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω. Τι θέσει έχετε να μου προσφέρετε. Δεν είναι μια κανονική δουλειά είναι μια δουλειά που είναι προϊόν της κοινωνίας μας όπου υπάρχει ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και όπου οι άντρε συνεχίζουν να νιώθουν ότι μπορούν να αγοράσουν σεξουαλικέ υπηρεσίε από τις γυναίκες. Το σουηδικό μοντέλο μειώνει τη ζήτηση και στη Γαλλία είδαμε ότι επιτέλους σε όλη την Ευρώπη αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι πορνεία και αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράση κατά της. Προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι 12 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και η Επιτροπή θα ψηφίσει στις 23 Ιανουαρίου και ε, θα πάει στην δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Μπορούμε λοιπόν τώρα να αφήσουμε το σημείο 7 και να προχωρήσουμε στο σημείο 8 εξάλληψη των βασανιστήριων στον κόσμο και δίνω το λόγο στην ε, συντάκτρια την κυρία Γιανακουδάκη. Thank you. And I'd like to... Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις ευρωβουλευτές που έμειναν μέχρι το πικρό τέλος, κυρίως την Μάριον που έχει να πιάσει το τρένο ε, να πάρει το τρένο. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη γιατί νομίζω ότι έχουν σβήσει και τη θέρμανση εδώ μέσα εκρίζωση των βασανιστήριων στον κόσμο υπό την οπτική του φίλου. Εστιάζω λοιπόν την προσοχή στις γυναίκες. Υπάρχουν ατέλειωτοι κατάλογοι βασανιστήριων όταν μιλάμε για τον ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων, καταναγκαστική γάμη, δολοφονίες, ε, στήρωση, ένα σωρό ε, τα έχω πει όλα όσα μπορούσα με δεδομένο του περιορισμένου αριθμού ε, λέξεων. Ε, μπορούμε να τα περιλάβουμε όσα, δεν, όσα έχω ξεχάσει ε, ή παραλείψει ε, με τροπολογίες. Δυστυχώς τα βασανιστήρια αυξάνονται και φαίνεται ο κόσμος να, ότι ο κόσμος βρίσκει όλο ένα και περισσότερους τρόπους για να βασανίζει. ελπίζω πως όλοι λοιπόν θα συμβάλλετε με τροπολογίες, οπότε θα αφήσω τους συναδέλφους να μου πούν τα σχόλιά τους τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμσεν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια η οποία έφτιαξε μια πολύ καλή γνωμοδότηση που νομίζω θα ενισχύσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην έκθεση. Με αυτή την ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τονίζεται ο λιθοβολισμός, ο κροτηριασμός των γεννητικών οργάνων, κατοίκων βία, καταναγκαστική γάμη και ένα σωρό άλλα που θα πρέπει να θεωρηθούν ως μορφές βασανιστήριων. <coughs> και προτείνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα λαμβάνει αυτά υπόψη σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στην αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει καθώς και στο διάλογο με τις τέτοιες χώρες. Ε, είναι μορφές ε, βασανιστήριων ε, όπως ε, ο ακροτηριασμός των γενετικό, γυναικείων γενετικών οργάνων. Όλοι ξέρουμε τις φρικτές επιπτώσεις αυτού, αυτού και θα πρέπει να το λέμε όπως είναι. Είναι βασανιστήριο. Η κατοίκον βία είναι επίσης ένα ευρύ εκτεταμένο πρόβλημα. Πολλές γυναίκες προκινδυνεύουν να πέσουν θύματα ε, κατοίκων ε, βίας, ε, ε, καρκίνου και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Επίσης θα πρέπει να θεωρήσουμε ως βάρβαρο τρόπο εκτέλεσης τον λιθοβολισμό. Δεν θα έπρεπε να κάνει να υφίσταται σήμερα ημέρα. Έπειτα, η ομάδα των ομοφιλόφιλων είναι πολύ ευαίσθητη ομάδα, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι προτάσεις λοιπόν της εισηγήτριας είναι σημαντικές, ε, είναι σύμμορφες με τις διεθνείς συμβάσεις περί γυναικείων δικαιωμάτων και στηρίζω την πρόταση για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Γιανακουδάκη, θέλετε να πάρετε το λόγο για να κλείσετε, παρακαλώ. Α, όχι, θα τα πω στα σουηδικά κι εγώ αυτά που έχω να κάνω παρατηρήσει. Κύριε Γιανακουδάκη, παρακαλώ, γρήγορα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ γιατί θα πάρω εγώ ο ίδιο τον λόγο τώρα ε, γιατί είμαι σκιώδη, εισηγητή. Σα ευχαριστώ για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότηση, γιατί αναφέρετε όλα τα θέματα που έπρεπε εδώ να αναφερθούν. Μιλήσατε για τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και της εκμετάλλευσης καλύψατε όλα τα πιο σημαντικά ζητήματα εδώ. Ε, ίσως θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες ε, σε σχέση με το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ και το 1889 που αφορούν και υπογραμμίζουν τη σημασία της βελτίωσης της ε, παιδείας αλλά και της ε, συνειδητοποίησης όλων αυτών των προβλημάτων ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντικό η UNICEF και η UN Women είναι, ε, δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο λήψη αποφάσεων να έχουμε περισσότερη ισότητα των φίλων, γιατί πολλοί άντρε είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν τι αποφάσει συνήθω και αν θέλουμε να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα πρέπει να έχουμε περισσότερε γυναίκε που αντιπροσωπεύουν τις γυναίκες στα όργανα λήψης αποφάσεων. Επίσης, νομίζω πως είναι καλή ιδέα να πούμε δύο λόγια για την Διεθνή Σύμβαση Γυναικών. Κάπως να το προσθέσουμε και αυτό. Και πάντως σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ καλή γνωμοδότηση, την πολύ καλή πρότασή σας και θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και εγώ και τώρα έχετε εσείς το λόγο. ευχαριστώ. Δεν θα αντισταθώ. Νομίζω πως ε, οι διερμηνές ήταν ε, τέλεια. Θα το χρησιμοποιήσω και στο, στο μανιφέστο μου ότι η Γκου αρχίζει να λέει πως είναι εξαιρετική συντηρητική. Όχι, το έλεγα για τη διερμηνέα. Ε, Θα βάλω και εγώ κάποιες ε, τροπολογίες γιατί ήταν λίγες οι λέξεις. Ε, ναι, ναι, επιτέλους μιλάμε και σοβαρά για τους ε, διερμηνείς. Και τώρα θα τα πω πάλι σου ειδικά. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Προθεσμία υποβολής τρυπολογιών 13 Δεκεμβρίου στις 12. Η Επιτροπή θα ψηφίσει 22-23 Ιανουαρίου του 2014. Η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει 10 Φεβρουαρίου. Και στην Ολομέλεια του Μαρτίου θα συζητηθεί. Και έτσι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να περάσουμε στο 9 διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα, περνάμε στο 10 που είναι η επόμενη συνεδρία η οποία θα πραγματοποιηθεί 16 Δεκεμβρίου 3 με 6.30 εδώ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ και κλείνουμε μία ώρα και έξι λεπτά πριν την ώρα μας. Tack så hemskt mycket till alla eh, tolkar. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς.